Okay, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σας καλωσορίζω στο επόμενο θέμα της σημερινής συνεδριασής μας. Θα δούμε μαζί τα σημεία 17 και 18 σε συνεργασία με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Καλωσορίζω και τον πρόεδρο της Επιτροπής αυτής. Μετά την άφετη, ίσως η καλύτερη επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπέρτ Λάγκε είναι εδώ μαζί μας ο συνάδελφός μου από την κάτω Σαξονία. Σας καλωσορίζω όλους λοιπόν. Σημείο 17. Στρατηγικές για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Η πρώτη εξέταση της έκθεσης Ιδίας Πρωτοβουλίας της ΑΦΕΤ για τις σχέσεις Ευρώπης-Κίνας ε, βρίσκεται στη σημερινή μας ε, ημερήσια διάταξη, αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε αυτή τη δημόσια ακρόαση με το ίδιο θέμα σε συνεργασία, όπως είπαμε, με την Επιτροπή Ίντα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας. Έχω μαζί, μου, έχω μαζί μου δίπλα μου τον κύριο Γιάν Βάιντενφίλτ, που είναι επικεφαλής του, της μονάδας ε, πολιτικής για την Κίνα στο Ινστιτούτο Μερκατόρ στο Βερολίνο. Έχουμε μαζί μας επίσης τον κύριο Φραντς Φαντερ Πούτερ, που είναι ερευνητής στο Ινστιτούτο Κλίνγκεντέλ στη Χάγη και μέσω συνδέσμου τηλεδιάσκεψης με το Πεκίνο. Έχουμε μαζί μας τον ε, κύριο Ματς Χάρμπον που είναι πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα από το Πεκίνο. Δεν ξέρω αν μας ακούει, μάλλον όχι όμως. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη σύνδεση. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στα βασικότερα ζητήματα που σχετίζονται με τις ε, σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας θα μιλήσει ε, πρώτα ο κύριος Βάιντενφελ για τη στρατηγική της Κίνας στην Ευρώπη και θα μας ε, κάνει κάποιες προτάσεις για το πώς θα διαμορφωθεί η δική μας ε, απάντηση στη στρατηγική της Κίνας. Δέκα λεπτά έχετε και στη συνέχεια ο κύριος Πούτεν, Πούτεν θα μας μιλήσει για τη θέση της Κίνας στο μελλοντικό παγκόσμιο γίγνεσθε και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Χάρμπον. Ε, παρακαλώ κύριε Βάιντενφελ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ ε, σε αυτήν την καλύτερη ε, από όλες τις ε, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και δεν είναι βεβαίω ε, υπερβολή να πει κανεί ότι έχουμε νέα στοιχεία στι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα. Και ε, ένα από τα πιο δύσκολα στοιχεία ε, είναι ότι δυστυχώς η Κίνα δεν φαίνεται να συγκλίνει με τα φιλελεύθερα οικονομικά και πολιτικά πρότυπα. Τα τελευταία δέκα χρόνια είχαμε τέτοια δείγματα, αλλά του τελευταίους 12 μήνες ιδιαιτέρω φαίνεται ότι πραγματικά η Κίνα ακολουθεί έναν δικό τη δρόμο. Αυτό βεβαίω θα δημιουργήσει προστριβέ, αναπόφευκτα, στις σχέσεις μας ε, και θα μας φέρει ακόμη και αντιμέτωπους ε, στο μέλλον. Το γεγονό ότι με προσκαλέσατε να μιλήσω σήμερα για τι στρατηγικέ τη Κίνα ε, στην Ευρώπη αφορά και ένα νέο στοιχείο. Η Κίνα ε, έχει μεγαλύτερη παρουσία στην Ευρώπη, οικονομικά, πολιτικά ή ακόμη και ως φορές ασφάλειας από ποτέ. Να δούμε λίγο τις οικονομικές δραστηριότητες της Κίνας, καταρχάς, στην Ευρώπη. Sorry about that. Λοιπόν, τα καταφέραμε να δούμε λίγο τις ε, οικονομικέ δραστηριότητε τη Κίνα στην Ευρώπη. Τα, τα εξωστρεφή στοιχεία ε, τη ε, Κίνα, της Κίνας, της βιομηχανικής πολιτικής της Κίνας, όπως το Made in China 2025, αλλά και οι στρατηγικέ επενδύσεις κρατικών επιχειρήσεων τη Κίνα στην Ευρώπη, θα συνεχίσουν να αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Και παρά το γεγονό ότι καθορίστηκε ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις εξωστρεφείς άμεσες ξένες επενδύσεις, που έχει ως στόχο να περιορίσει την εκροή κεφαλαίων. Δεν υπάρχει κανένα δείγμα που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στην ανωδική πορεία των ε, κινέζικων επενδύσεων στην Ευρώπη. Ε, με δεδομένο ότι προετοιμάζονται συμφωνίες αξίας 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπάρχει σταθερό έδαφος για κινέζικες αξίες στην Ευρώπη το 2018. Υπάρχει μια τέτοια ανωδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το μέγεθος λοιπόν των ε, κινέζικων αξέ στην Ευρώπη δεν είναι πρόκληση από μόνο του. Όμως οι στόχοι και οι πηγές αυτών των επενδύσεων αποτελούν πηγή ανησυχία. Στα τελευταία χρόνια το μεγαλύτερο μερίδιο των ε, κινέζικων αξέ στην Ευρώπη κατευθύνθηκαν στι μεταφορές, τις υπηρεσίες κοινή ωφέλεια και τι υποδομέ που είναι κλάδοι που συνδέονται και με την εθνική ασφάλεια. Ενώ οι τομείς υψηλής τεχνολογίας και προηγμένης μεταποίηση που αποτελούν κέντρο βεβαίως του σημερινού και του μελλοντικού πλούτου των εθνών ε, αποτελούν επίσης στόχο των κινέζικων επενδύσεων. Το γεγονός βεβαίως ότι οι επενδύσεις αυτές γίνονται από κρατικά σε επιχειρήσεις της Κίνας επίσης είναι ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο. Ε, προτάσεις που συζητούνται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την δημιουργία ενός μηχανισμού ελέγχου των ε, επενδύσεων στην Ευρώπη αποτελούν ένα, ένα σημαντικό βήμα. Ωστόσο, ε, στην καλύτερη περίπτωση αυτό θα μπορούσε να είναι μια βραχυπρόθεσμη αντιστάθμιση των κινδύνων η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να μεταρρυθμίσει εν γέννη την πολιτική ανταγωνισμού της. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που σχετίζεται με τα εξωστρεφή στοιχεία της ε, εξωτερικής ε, και εμπορικής πολιτικής της ε, Κίνας θα είναι η απάντηση που θα δοθεί από πλευράς Ευρώπης σε ζητήματα ή θέματα όπως το 5G, το ίντερνετ των πραγμάτων και η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, ε, γίνεται όλο ένα και πιο ορατή η πολιτική επιρροή της Κίνας στην Ευρώπη και παρό το γεγονός ότι συνήθως βλέπουμε ρωσικές αντίστοιχες ε, δράσεις, υπάρχουν σημαντικοί λόγοι να πιστέψει, για να πιστέψει κανείς ότι και η Κίνα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση μέσω μακροπρόθεσμα. Και ε, το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα ε, καταβάλει συστηματικές προσπάθειες προκειμένου να επανακαθορίσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο οι Ευρωπαίοι βλέπουν την πολιτική και οικονομική παρουσία της Κίνας στην Ευρώπη και του Πεκίνου εν γέννη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, υπάρχουν λοιπόν προσπάθειες ε, οι οποίες προσπαθούν να διαμορφώσουν και να σκιαγραφίσουν την παρουσία της Κίνας με θετικότερα χρώματα αλλά και να, κάνουν, να φημώσουν κριτικές ε, ε, φωνές. Και το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά φαίνεται η Κίνα και το κομμουνιστικό της κόμμα να θεωρούν ότι το δικό του σύστημα είναι ανώτερο από εκείνο της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Μάλιστα γίνονται και συγκεκριμένες προσπάθειες ώστε να καταστεί ακόμη πιο δημοφιλές στον υπόλοιπο κόσμο το κινέζικο μοντέλο. Επειδή δεν έχω πολύ χρόνο για να μιλήσω με λεπτομέρειες για τα εργαλεία επιρροής που χρησιμοποιεί η Κίνα, θέλω να σας δώσω ένα βασικό μήνυμα. Η Κίνα ήδη αξιοποιεί και μετέρχεται μια σειρά από προηγμένα εργαλεία επηρεασμού της κοινή γνώμης στην Ευρώπη που κατευθύνονται κατά κύριο λόγο στις πολιτικές και επιχειρηματικές ελίτ, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Το γεγονό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα χρησιμοποιεί βεβαίω αυτά τα εργαλεία δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα έχουν αντίκτυπο, αλλά υπάρχουν κάποιε εξελίξει που μα ε, οδηγούν σε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να σταθεί με συνέπεια και ενότητα απέναντι στην Κίνα. Ε, σε ζητήματα όπως είναι η ε, υποχρεωτική και απαραίτητη τήρηση του κράτους δικαίου στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας λοιπόν έχει ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία και στα ΜΜΕ στην Ευρώπη αλλά και σε δεξαμενές σκέψεις και στα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Η επιτυχής λοιπόν αντιμετώπιση των κοινοζικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη ε, θα συμπεριλάβει αναγκαστικά ε, επενδύσεις ε, σε δεξαμενές, πλοίο, ε, δεξαμενές σκέψεις και πανεπιστήμια και την διαπαιδαγώγηση βεβαίως και της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης σχετικά με τη φύση αυτών των προσπαθειών που καταβάλει η Κίνα για, τον, για την επιρροή προς όφελός της της ευρωπαϊκής κοινή γνώμης. Συμπερασματικά θα ήθελα να επισημάνω επίσης ότι υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια ως προς την ε, παρουσία της Κίνας στην Ευρώπη. Η ε, παρουσία της Κίνας λοιπόν ε, είναι ολοένα και μεγαλύτερη σε τρίτες χώρες και ιδίως στην Ευρώπη. Δύο είναι τα βασικότερα παραδείγματα. Πέρσι το ναυτικό της Κίνας συμμετείχε σε κοινή στρατιωτική εκπαίδευση με την άσκηση μάλλον με τη Ρωσία στη Βαλτική θάλασσα. Την ακριβώς προηγούμενη χρονιά είχε γίνει μια αντίστοιχη στρατιωτική επιχείρηση στη Μεσόγειο και Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τους τελευταίους 12 μήνες ένα μέλος του ΝΑΤΟ, η Τουρκία, φλερτάρει με την ιδέα να ε, ενταχθεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Αγκάρης Και παρά το γεγονός ότι η Κίνα προς το παρόν τουλάχιστον δεν επιθυμεί ε, ευθεία αντιπαράθεση με τον ΝΑΤΟ, φυσικά καθόλου δεν τη δυσαρεστεί αυτή η εξέλιξη με τον Ερντογάν. Και αυτό αυτό ίσω είναι και ενδεικτικό της διαβρωτικής ε, στάσης εν γέννη της Κίνας απέναντι στον ΝΑΤΟ. Βεβαίως, η παγκόσμια πολιτική ασφάλεια τη Κίνα πρέπει να μας απασχολήσει εδώ στην Ευρώπη. Χρειάζεται μεγαλύτερο έλεγχο, μεγαλύτερη επαγρύπνηση από τους Ευρωπαίους πολιτικούς, ε, πέρα από την καθαρά οικονομική λοιπόν και πολιτική δραστηριοποίηση της Κίνας ε, στην Ευρώπη και θα ήθελα πολύ να συζητήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερος ομιλητής, ο κ. Φάντερ Πούτεν, ε, θα μας μιλήσει για το μέλλον της ε, Κίνας, την εξωτερική πολιτική ε, ασφάλειας της Κίνας θεωρήσεις του, μέλλον, του μελλοντικού ρόλου της Κίνας ε, της, στη διεθνή πολιτική είναι ο τίτλος. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά γι' αυτό θα σας μιλήσω. Δεν θέλω να προβλέψουμε το ρόλο της Κίνας, αλλά να φράσω κάποιες σκέψεις, να εστιάσω κάποια στοιχεία για τα οράματα της Κίνας, αυτά που έχει ήδη παρουσιάσει η Κίνα, για το δικό της μελλοντικό ρόλο στη διεθνή πολιτική και με έναν τρόπο που θα δείχνει και τη δική μου προσωπική ερμηνεία αυτών των οραμάτων. Η κινέζικη ηγεσία και ιδιαίτερος ο πρόεδρος πολύ συχνά αναφέρεται στην ανανέωση, ε, αναζωογόνηση. Σε πολλές ομιλίες του έχει πει, για παράδειγμα, ότι σχετίζεται με το γεγονός ότι η Κίνα είχε μείνει πίσω, ήταν οπισθοδρομική στο παρελθόν, κάτι που είχε καταστήσει την χώρα ευθραυστή, ευαίσθητη και ότι η ανάπτυξη την κάνει ε, δυνατή. Η αναζωογόνηση είναι το πιο σημαντικό όνειρο του κινέζικου λαού, λέει ο πρόεδρος. Ότι η χώρα θεωρεί, πρέπει να το θεωρεί ως βασικό της στόχο. Αναφέρεται στην ιστορία της ε, Κίνας, όπου ήταν, ε, η Κίνα ήταν αδύναμη, ε, ήταν ευάλωτη. Πολλά πράγματα είχαν συμβεί εκείνη την εποχή. Ο πόλεμος του οποίου που τελείωσε το 1842 για παράδειγμα ορισμένες από τις σημαντικές ε, αλλαγές ε, τα σημαντικά γεγονότα τα οποία εξέθεσαν την, το, το πόσο ε, ευάλωτη ήταν η χώρα ήταν η απώλεια της αυτονομίας της η απώλεια ε, επικράτεια στο Χογκόν και Ταϊβάν ε, έχασε τη θέση της ως ε, μεγαλύτερη οικονομία και ως ηγέτης σε περιφερειακό επίπεδο. Όμως η Κίνα ανέκτησε την αυτονομία της, ανέκτησε το Χονγκ Κόνγκ, δεν τα κατάφερε ακόμα, δεν τα έχει καταφέρει ακόμα να γίνει η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, είναι η δεύτερη αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καταφέρει ακόμα να περάσει τον έλεγχο της Ταϊβάν και ακόμα δεν είναι ηγέτη αδύναμη στην περιφερειακή πολιτική της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ε, μιλάει λοιπόν για εθνική αναζωογόνηση ο πρόεδρος, αλλά αυτό που κυρίως εννοεί κατά την άποψή μου είναι η ανάκτηση αυτών των τεσσάρων στοιχείων. Ένα άλλο πολύ σημαντικό κομμάτι της θέσης της Κίνας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τις διεθνείς σχέσεις. Βλέπετε εδώ ε, μια άλλη ρίστη πίνγκ από το 2013. Την έχει επαναλάβει άλλωστε λέει ότι η Κίνα θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα όλων των χωρών να επιλέξουν ανεξάρτητα το κοινωνικό του σύστημα και το, την οδό της ανάπτυξής τους. Ανεξάρτητα αν είναι μικρές ή μεγάλες, λέει, οι χώρες είναι ίσα ισότιμα μέλη της διεθνούς κοινότητας. Ανεξάρτητα το πόσο μεγάλες ή μικρές είναι, πόσο ισχυρές ή αδύναμες. Εδώ έχουμε δύο πτυχές. Πρώτον, την πολιτιστική ποικιλία, κάτι που προωθεί η Κίνα ποσο ισχυρες οι αδυναμες εδω εχουμε δυο πτυχες πρωτον την πολιτιστικη ποικιλια κατι που προωθει η κινα εδω και αρκετό καιρό, ότι ε, ενδεχομένως θα μπορούσε να ερμηνευθεί όσο ότι δεν υπάρχουν καθολικές παγκόσμιες αξίες. Κάθε χώρα θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει το δικό της πολιτικό και οικονομικό σύστημα. Οπότε οι φιλελεύθερες πολιτικές και οικονομικές αξίες που προωθούν οι δυτικές χώρες ως καθολικές αξίες ε, δεν είναι τέτοιες. Το άλλο που προκύπτει από αυτό που είπε ο πρόεδρος είναι ότι στη διεθνή διπλωματία όλοι είναι ίσοι και δεν υπάρχουν προνομιούχες ε, δυνάμεις. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να υποσκάψει το παραδοσιακό ρόλο κάποιων δυτικών κυρίως δημοκρατιών ε, στη διεθνή διπλωματία. Οι δυτικές δυνάμεις αλλά και οι η Ιαπωνία, τελευταία και η Ρωσία έχουν για την Κίνα προνομιακές, ε, προνομιακές θέσεις που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Ο Τέγκ Σιαοπίνγκ τώρα είχε πει αυτό που αναφέρει η συγκεκριμένη διαφάνεια το 1974 να μιλώντας στη, συνέλευση, Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ε, είχε πει Βέβαια πολλά από αυτά που έλεγε τότε δεν ισχύουν πλέον, αλλά ορισμένα ε, παίζουν ακόμα σημαντικό ρόλο στο όραμα της Κίνας για το μέλλον. Τότε ο Τέν Σιαοπίνγκ είχε πει ότι η Κίνα έχει μια ευθύνη να δρά ε, εξ και εκ μέρους των αδύναμων και καταπιεσμένων του, όλου του κόσμου εναντίον των καταπιεστών των χωρών που τους καταπιέζουν τότε ήταν οι Ηνωμένες και η Σοβιετική Ένωση σύμφωνα με την λογική της Κίνας. Είχε πει επίσης ότι η Κίνα δεν είναι υπερδύναμη ούτε και θα γίνει ποτέ όπως για παράδειγμα η Σοβιετική Ένωση ή οι Ηνωμένες Πολιτείες εκείνη την εποχή. Η, η Κίνα εξακολουθεί να τις θεωρεί βέβαια υπερδυνάμεις ακόμα. Τώρα, ε, για να καταλάβετε τα προηγούμενα, έχω εδώ ένα χρονοδιάγραμμα, μια γραμμή χρόνου. Η Κίνα έγινε παγκόσμιος πολιτικός παίκτη από το 1917 όταν κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Δηλαδή έναν αιώνα πριν. Ε, έγινε μέλος της ε, ε των Εθνών ε, το 19 και μόνιμο μέλος του, της Συμβουλής Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, το 1945. Πάνε πολλά χρόνια από τότε. Μετά το 1945 λοιπόν, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισε να αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγάλες δυνάμεις στον κόσμο και από τότε εστίαζε όλο και περισσότερο στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Το 1974 ο Τέκ Τζιαοπίνγκ ε, κάνει αυτήν την ομιλία από την οποία σας διάβασε ένα απόσπασμα. Πλέον παρουσιάζει τον εαυτό της ως άτυπος ηγέτης ε, του αναπτυσσόμενου κόσμου του G77 και το 2013 ε, παρουσίασε και την ε, πρωτοβουλία ε, Belt and Road ε, της ζώνης και του δρόμου. δηλώνοντας ότι η προσέγγιση του δυτικού κόσμου δεν ήταν σωστή και τώρα πλέον θα πρέπει η Κίνα να λάβει την, τον κυρίαρχο λόγο της οικονομικής ανάπτυξης ε, παγκοσμίως. Τέλος, ε, βλέπετε εδώ ε, ένα χρονοδιάγραμμα για, την, ε- για τον υπόλοιπο αιώνα, τις επόμενες δεκαετίες. Το 2021 το σχέδιο είναι να είναι σχετικά ευημερούσα χώρα, το 2035 να είναι παγκόσμια ηγέτη στην καινοτομία και το 2049 να είναι παγκόσμιος ηγέτης σε ό,τι αφορά την πολιτική επιρροή που θα έχει. ο Σι Τζιμπίνγκ, ο πρόεδρος, θεωρεί ότι μέχρι το 2049 ε, η Κίνα θα έχει πετύχει το εθνικό της στόχο για εθνική αναγέννηση ή ε, αναζωογόνηση. Η, η Κίνα ε, με συνέπεια εργάζεται στο, προς την κατεύθυνση της μείωσης της διαφοράς που τη του χάσματος που τη χωρίζει ανάμεσα στην στην, με, από τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, ε, από τις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης. Επίσης θέλει να βοηθήσει και τις άλλες αναπτυσσόμενες χώρες να κάνουν το ίδιο, βοηθώντας τις οικονομικά, αλλά και αντισταθμίζοντας την οικονομική και πολιτική επιρροή της Δύσης στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Δεύτερον, η Κίνα ε, εργάζεται προκειμένου να δώσει τέλος στον πρωταρχικό κυριαρχικό ρόλο της, ε, των ΗΠΑ στην Ασία ε, προσπαθεί να ξεπεράσει τις ΗΠΑ και οικονομικά και διπλωματικά και τεχνολογικά. Τρίτον, η Κίνα θέτει τον εαυτό της ως πρώτο μεταξύ ίσων μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και μεταξύ των ε, μεγάλων δυνάμεων του κόσμου. Τέταρτον, προσπαθεί να διατηρήσει την τρέχουσα παγκόσμια ε, αρχιτεκτονική διακυβέρνησης, αφαιρώντας όμως τον ηγετικό ρόλο της δύση και τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι φιλελεύθερες αρχές. Τέλος για την ευρωπαϊκή στρατηγική, να κάνω την εξή παρατήρηση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσει με την Κίνα για θέματα ανάπτυξης, γιατί για την Κίνα η ανάπτυξη είναι εξαιρετικά σημαντική ε, και για την, ε, για την νομιμοποίηση του δικού της ρόλου στον κόσμο. Η Κίνα έχει να παίξει ρόλο στην διεθνή παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι η Κίνα προσπαθεί να δημιουργήσει μια ένταση, μια ε, τριβή ανάμεσα στις αναψιόμενες χώρες και τη Δύση και προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίβαρο στις νομές Πολιτείες. Τέλος, υπάρχει το θέμα των αρχών. Ο Γιάνν Βάιντενφελτ το έθιξε. Η Κίνα δεν, την Κίνα δεν την ενδιαφέρουν οι δυτικέ φιλελεύθερε αρχέ που είναι σημαντικέ και για την Ευρώπη. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη. Okay, thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Φαντπούτεν. Οι Βρυξέλλες καλούν. Έχουμε σύνδεση με το Πεκίνο. Ah Hello Hello Hello Oui. Attends, Can you hear me now Με ναι, ακούτε Να σας ακούω. Α, τι ωραία. Σας καλούμε την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Συνεδριάζουμε την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Και είστε ο τρίτος ομιλητής τώρα. Και μας είπαν ότι έχετε μια εισήγηση να κάνετε σχέση με τον επικοδομητικό διάλογο. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Λέγομαι Μάτς ε, Χαμπορν, πρόεδρος του Επιμελητήριου της Ένωση στην Κίνα. Εμείς θεωρούμε ότι τώρα πια σε σχέση με το εμπόριο και τι επενδύσει είναι η σειρά τη Κίνα. Η Κίνα θα πρέπει βεβαίω να τηρήσει κάποιε δεσμεύσει σε σχέση με ανοίγματα. His recent speech in Bao was followed by more concrete announcements. And European businesses, we expect more in 2018, the year when China celebrates the 40th anniversary of the open door policy. We have a basic assumption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 Ευχαριστώ πάρα πολύ το Πεκίνο. Συνάδελφοι, ακούσαμε τις τρεις εισηγήσει. Έχουμε περίπου ένα μισάωρο για συζήτηση με τους εισηγητέ μας. Ο Μπερλάνκε πρώτα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σκέφτομαι ότι ναι, πολλές από τις θέσεις που έχουμε συζητήσει είναι αμυντικές, είναι αμυντικογενείς. Λέμε ότι η Κίνα κάνει το τάδε, το δίνα, προσπαθεί να πετύχει περισσότερη πολιτική επιρροή κλπ. Και αυτό σχετίζεται και με την αδυναμία των ευρωπαϊκών πολιτικών και ιδιαίτερα με την αδυναμία να μην έχουμε μια πραγματική βιομηχανική στρατηγική. Εντάξει, οι Κινέζοι έχουν τη δική του στρατηγική. Η δικιά μας όμως ποια είναι. Ποια είναι η στάση μας σε αυτά τα θέματα πολιτικής. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ισορροπία λοιπόν. Εντάξει, στο εμπόριο υπάρχουν διάφορα προβλήματα, τα ακούσαμε, ποια είναι, υπάρχει άνηση μεταχείριση σε σχέση με τις κρατικές επιχειρήσεις, υπάρχουν προβλήματα σε επενδύσεις και είναι σημαντικό βεβαίως να βρούμε κοινό έδαφος με τις κινέζικες αρχές για συμφωνίες επενδυτικές που τώρα διαπραγματεύονται νομίζω 17 και μετά το 19ο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος νομίζω ότι είναι πιο διαθέσιμη για συμφωνίες. Έχουμε και το θέμα της σταθεροποίησης των πολυμερών εμπορικών συστημάτων και της συνεργασίας στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. και δηλώσεις κατά προστατευτικών μέτρων. Εκτός λοιπόν από την κριτική και τι επικρίσει για τι πρακτικές στην Κίνα θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παγκοσμίω χρειαζόμαστε την Κίνα ως εταίρο στα πλαίσια του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτή είναι η απόψή μου, αλλά είναι και ένα ερώτημα αυτό ταυτόχρονα προς τους εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Θα προτείνω να ακούσουμε κάποια σχόλια από τους συναδέλφους και μετά θα απαντήσουν οι συγγητές. Φασμπέλντερ, ο συγγητής είναι ο επόμενος ομιλητής. Βας Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δεν περιμένω αυτό τόσο γρήγορα η σειρά μου, αλλά τέλος πάντων. Ακούσαμε πολλά ενδιαφέροντα σήμερα το απόγευμα. Και για μένα ως εισηγητή αυτά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον που άκουσα. Και άκουσα με ενδιαφέρον επίση τα συγκεκριμένα στοιχεία σε σχέση με την ανάπτυξη και την εξέλιξη της Κίνας, η οποία είναι όλο και πιο διεισδυτική στην Ευρώπη. Να πω το εξή σύντομα. Ένας ε, γνωστός καθηγητής, υπεύθυνο, μάλλον καθηγητής ε, κινέζικων σπουδών, συνικών σπουδών στην Ευρώπη, έλεγε παλιά ότι οι Κινέζοι έχουν στρατηγική, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει. Οπότε στρέφουμε προς τους προσκεκλημένους μας. Κύριε Φαντεμπούτεν, το αναφέρατε στην εισήγησή σας. μήπω λοιπόν έχει έρθει η ώρα επιτέλου και η Ευρώπη να χαράξει μια δικιά της στρατηγική, γιατί έχουμε σημειώσει μεγάλη καθυστέρηση. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι οι Κινέζοι εποφελούνται κάθε δικής μας αδυναμίας και την εκμεταλλεύονται αμήλικτα υπέρ τους. Οπότε πρέπει να επαγρυπνούμε. Τι γίνεται λοιπόν με τη στρατηγική, τη συνολική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Κίνα. Το να εκμεταλλευόμαστε τις ανεμίες των άλλων πως ε, κάνει η Κίνα και η έλλειψη στρατηγικής εκ μέρους της Ένωσης ε, είναι μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Οπότε θα ήθελα την άποψή σας. Και ακούσαμε προηγουμένως ότι οι δικές μας φιλελεύθερες αξίες δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν αλλά βλέπουμε ότι ταυτόχρονα έχουν μια δημόσια διπλωματία οι Κινέζοι παγκοσμίω, κάνοντα έκκληση για αύξηση των επενδύσεων εκεί. Και πριν από δύο χρόνια η αντιπροσωπεία της Ένωσης στο Πεκίνο μου είχε πει ότι έχει φτάσει η ώρα πια για να γίνουν μελέτες ανεξάρτητες από τα πολιτικά κόμματα σε σχέση με την πολιτική προσέλκυση επενδύσεων στην Κίνα. Τι γίνεται με αυτό. Ο λόγο τώρα στο Γιολάινερ, που είναι πρόεδρο τη αντιπροσωπεία για τη σχέση με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, έχουμε έναν ανταγωνισμό των συστημάτων που εμφανίζεται στο προσκήνιο και από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί για πολλά χρόνια. Άλλωστε, ε, ακούστηκε ότι ο Xi Jinping έχει σχέδιο έως το 2049. Το κινέζικο όνειρο λοιπόν αυτό θα εκπληρωθεί έως τα μέσα του αιώνα. Είπατε το 2035 θέλει να είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη παγκοσμίω και το 2049 και η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στον κόσμο. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόκληση την οποία δεν, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε γιατί τα συστήματα είναι πολύ διαφορετικά. Εμείς έχουμε την φιλελεύθερη δημοκρατία, εκεί υπάρχει ένα αυτερχικό καθεστώς, το οποίο εξυγχρονίζεται βεβαίως και που μάλιστα προσφέρεται πλέον ως μοντέλο, ως υπόδειγμα και για άλλες χώρες στον κόσμο. Ε, νομίζω ότι υπάρχει αντίκτυπος αυτής της κινέζικης παρουσίας ήδη στον υπόλοιπο κόσμο, σε άλλες χώρες. Δεν θα έλεγα απαραίτητα ο κύριος Όρμπαν, αλλά ο κύριος Ερντογάν σίγουρα ε, στον έναν ή στον άλλο βαθμό μιμείται ε, το κινέζικο μοντέλο. Ο Μπέρντ Λάγκε άλλωστε έθεσε το θέμα στις σωστές του βάσεις. Εμείς τι κάνουμε είναι το ερώτημα. Πώς θα καταστήσουμε το ευρωπαϊκό υπόδειγμα πιο ελκυστικό. Πώς ε, θα το παρουσιάσουμε ενδεχομένως και με μια νέα ορμή, με μια νέα δυναμική στον υπόλοιπο κόσμο. βεβαίως πέρα από τις αξίες μας ε, πρέπει να εξυπηρετήσουμε και τα οικονομικά μας συμφέροντα. Και εκεί η Κίνα πράγματι έχει προβάδισμα στις υποδοσμές, ε, στην βιομηχανία. Πρέπει σίγουρα να δούμε τι θα κάνουμε αυτό το θέμα. Ε, είχαμε μέχρι τώρα μια φάση ανάκαμψης της οικονομίας στην Ευρώπη, αν και αρχίζουν και συσσωρεύονται σύννεφα στον ουρανό, ε, παρόλα αυτά το κρατούμενο που είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι ναι, είμαστε κατά του προστατευτισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως ότι δεν πρέπει να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας. Στον ανταγωνισμό λοιπόν υπάρχουν θέματα, δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Επίσης, ένα ακόμη θέμα ε, που μας απασχολεί και πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο είναι η παρουσία της Κίνας στο διαδίκτυο με τις εφαρμογές του και το λογισμικό του. Ε, πρόκειται για μια νέα, όπως την αποκαλούν πολλές πλευρές, ψηφιακή εποχή που δεν ξέρουμε τι μας ε, επιφυλάσει. Συμπέρασμα λοιπόν ναι στη συνεργασία, αλλά με κριτικούς όρους και με κριτικό βλέμμα. Γιατί πολλοί νομίζω ότι εξακολουθούν να είναι θεροβάμονες και να ονειρεύονται κινέζικες όπερες, ε, έναν πολιτισμό 5.000 ετών, τον, ε, τις παγόδες. Όλα αυτά ωραία είναι, αλλά πρέπει κανείς να έχει ένα βλέμμα διεισδυτικό και να διαπιστώνει ακριβώς ποιες είναι οι εξελίξεις που τρέχουν. Αν θέλουμε πραγματικά να ζήσουμε και το, τα επόμενα χρόνια ε, με ειρήνη και συνεργασία. Τώρα ο, ο λόγος είναι της ΙΝΤΑ. Τον κύριο Βίνκλερ. Θα ήθελα να χαιρετήσω τον ε, Μάτς που είναι πρόεδρος ε, του ο μελητηρίου στην ε, Κίνα, ε, ένα τμήμα της έκθεσης μου στην Ίντα βασίζεται στις δικές του παρατηρήσεις. Είναι φυσικό αυτό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν, γιατί μιλάμε, έχουν άμεση ε, επαφή με τις επιχειρήσεις που, της Ευρωπαϊκής που ενεργοποιούνται, δραστηριοποιούνται στην Κίνα. Σήμερα αυτή τη στιγμή εισάγουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αγαθά αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων και εξάγουμε 1,5 δισεκατομμύριο ε, ε, προϊόντα αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Κίνα. αυτό είναι μόνο για τα αγαθά. Δεν μιλώ ούτε για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ούτε για τις υπηρεσίες, ούτε για τις επενδύσεις. Όταν λοιπόν λέμε ότι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας αντιμετωπίζουν κάποιες, κάποιες, κάποια καινούργια πραγματικότητα, νόμιζα ότι θα μιλούσατε για τον Αμερικανικό προστατευτισμό και τον κύριο Τραμπ. Δεν το κάνατε, αλλά και αυτό είναι ένα κομμάτι της καινούριας πραγματικότητας. Ο προστατευτισμός έρχεται, οποία έχει πληξεί από τις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή, από την Ουάσιγκτον. Οπότε πράγματι υπάρχουν καινούριε πραγματικότητε. Θα πρέπει να προσπιστούμε τα συμφέροντά μας και να τηρήσουμε τους κανόνες. Και ο πρόεδρος Xi Πιν και το Πεκίνο στις ομιλίες του αναλαμβάνει δεσμεύσεις που όμως ακόμα δεν έχουν υλοποιηθεί. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε απτά μέτρα όπως αυτά τα οποία έχουν, γίνει στα αυτοκίνητα, στο, στην αφηγική, στην, ε, ε, ε, στο, στον χρηματοοικονομικό τομέα κλπ. Και μιλούσαμε με τον Υφυπουργό Εμπορίου της Κίνας εδώ στις Βρυξέλλες χτες και συνάντησε και τον ε, Πίτροπο και τον κύριο Λάγκε και εμένα σήμερα και μιλήσαμε με ειλικρίνεια ότι θα πρέπει να επικρατήσει καλύτερη αλληλοκατανόηση και να είμαστε πιο ειλικρινεί στο διάλογό μας. Χρειαζόμαστε περισσότερο ειλικρίνεια και στον εσωτερικό μας διάλογο. Παράλληλα, με τις πολιτικές μας ε, πρόσβαση στις αγορές θα πρέπει να συζητήσουμε ποιοι είναι οι εσωτερικοί κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν και αν το 16 συν 1 πληρεί αυτούς τους κανόνες θα έπρεπε το 16 1 να γίνει ένα από τα στοιχεία της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ, λέει ο πρόεδρος. Περάμε στους υπόλοιπους ομιλητές που έχουν ζητήσει το λόγο. κυρία Ζούιτσα, Αντεκένε, Ζαραντήλ, Βάγγελ, Μπουτιχόφερ και ο κύριος Σόλτς. Ο κύριος Κούκαν. Θα κλείσω το κατάλογο των ομιλητών. Δύο λεπτά στον καθένα. Κύριε Σουίτσα, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, Πρόεδρε. Πράγματι, τα δύο συστήματα είναι ανταγωνιστικά. Ας μην το ξεχνάμε και ας μην ξεχνάμε ότι ε, ο πρόσκυνος μετά τους καινούριους κανόνες μπορεί να διατηρήσει την εξουσία απεριόριστα, χωρίς χρονικά όρια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς όμως το διάλογο με την Κίνα και να συνεργαζόμαστε επί τη βάση συγκεκριμένων κανόνων. Έχω την εξής ερώτηση. Μιλήσατε για το Χονγκ Κόνγκ και την Ταϊβάν. Είπατε ότι οι Κινέζοι επανέκτησαν το Χονγκ Κόνγκ αλλά όχι ακόμα την Ταϊβάν. Σε πρόσφατο ψήφισμά μας ε, επαναλάβαμε τη στήριξή μας στη συμμετοχή της Ταϊβάν στους διεθνείς οργανισμούς Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την Ταϊβάν. Γιατί όμως η Ταϊβάν δεν προσκληθεί ούτε πέρσι ούτε φέτος στην ε, διάσκεψη της Νοτιοανατολικής Ασίας και δεν συμμετέχει ούτε στο Μαγκόσμιο Οργανισμό Υγείας παρόλο που ε, είναι πάρα πολύ δραστήρια σε θέματα υγεία, δημόσιας υγείας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια Γι' αυτό η Κίνα θα πρέπει να σταματήσει να εμποδίζει την συμμετοχή της Ταϊβάν στους διεθνείς οργανισμούς γενικότερα. Θα είχατε να μας πείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριο Ζάραντι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχω την αίσθηση ότι ε, είμαστε μπερδεμένοι σε σχέση ε, με το πώς πρέπει να, χειριστούμε την, ε, την Κίνα. Είναι αντίπαλος, είναι εταίρος. Ε, νομίζω ότι ακόμη δεν έχουμε καταφέρει να χωνέψουμε τον, την αυξανόμενη επιρροή που έχει η Κίνα στο παγκόσμιο στερέωμα. Αν δείτε το χώρο, το, το, χάρτη, οι 20 ευρωπαϊκές χώρες ε, έχουν τη Γερμανία ως μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, ενώ η Γερμανία έχει ως μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της την Κίνα. Υπάρχει λοιπόν μια μεταστροφή ε, και αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει στο να χειριστούμε και να προσεγγίσουμε την Κίνα με ρεαλιστικότερους όρους ε, ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες διαφωνίες υπάρχει, υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής ε, τον οποίο, μπορούμε να, τον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε ανοιχτό διεθνές εμπόριο για παράδειγμα συγκεκριμένοι κανόνες μάλιστα Φαίνεται από τις παρουσιάσεις ότι η Κίνα προσπαθεί να επηρεάσει και τα πολιτικά πράγματα στην Ευρώπη, πανεπιστήμια, μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. κτλ. Προφανώς η Κίνα κάνει δημόσιες σχέσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, αλλά ας μην είμαστε υπερβολικά καχύποπτοι ούτε παρανοϊκοί με αυτά τα θέματα. Εγώ ε, διάβασα πρόσφατα στο Πολίτικο ένα άρθρο το οποίο αναφερόταν σε αυτή την πρωτοβουλία 16 συν 1 ως ένα σχέδιο της Κίνας για το πώς θα διαιρέσει και θα διχάσει την Ευρώπη. Νομίζω ότι χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα και νυφαλιότητα όταν εξετάζουμε αυτά τα θέματα. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Αν μην προσπαθήσουμε μόνοι μας να οικοδομήσουμε θεωρίες συνωμοσία και τέτοια πράγματα. Ας είμαστε ανοιχτοί, ας είμαστε ειλικρινείς, ας είμαστε ε, πρόθυμοι για συνεργασία και ρεαλιστές πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πολύ να σχολιάσω αυτό που είπατε για το 16 συν 1, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ λόγω της θέσης μου σήμερα. Ο κύριος Βάιγκελ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για τη δική μας στρατηγική απέναντι στην Κίνα. Και θα ήταν μεγάλο σφάλμα αν εξ αρχής θεωρήσουμε εχθρό ή αντίπαλο, ως εχθρό ή ως αντίπαλο την Κίνα ή ως ε, έναν, μια χώρα που μόνο κακό μπορεί να κάνει στα συμφέροντά μας. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στις επαφές μας με την Κίνα. Θέλω όμω να αναφερθώ σε ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Πρόσφατα έγινε μια συνδιάσκεψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά την περιφερειακή ασφάλεια στην ε, Νότια Κινέζικη θάλασσα και είχαμε μαζί μας μάλιστα διακεκριμένους εταίρους μας από την Ταϊβάν που συμμετείχαν στην ε, εν λόγω συζήτηση. Φυσικά για την Ταϊβάν οι πρόσφατες αλλαγές ε, που ήταν εν μέρη και δραματικές είχαν σοβαρό αντίκτυπο όσον αφορά τις ανησυχίες γύρω από τον τομέα της ασφάλειας της Ταϊβάν. Όταν η Ταϊβάν έχασε ε, σημαντικούς ε, αεροδιαδρόμους ε, γύρω από την επικράτειά της, πραγματικά ε, αυτό αποτέλεσε κίνδυνο για την αεροπορία και την ασφάλεια. Μάλιστα στην ε, διάρκεια του, του φόρουμ Μποάο που έγινε τον Απρίλιο ε, εισήλθε κινέζικο πλοίο στα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν ε, ως ε, επίδειξη δύναμης στρατιωτικής από την πλευρά της Κίνας. Και αυτά είναι ανησυχητικά. Παρ' όλα αυτά η Κίνα νομίζω ότι επικεντρώνεται κυρίως ε, στην εμπορική της πολιτική και επιδιώκει να εξασφαλίσει την ειρήνη και την ασφάλεια. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει μόνιμος ε, διάλογος μεταξύ Κίνας ε, και Ταϊβάν γιατί κάτι τέτοιο μόνο θετικά μπορεί να δράσει υπέρ της ε, ασφάλειας, της ε, συνολικότερης περιφέρειας της περιοχής αυτής ε, που περιλαμβάνει και την Κίνα και την Ταϊβάν. Ευχαριστώ κύριος Μπιρικόφερ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι καλή προσέγγιση. όπως μας είπε ένας από τους συζητητές να δούμε τι νέο υπάρχει. Ποια τα νέα στοιχεία όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο μερών, Ευρωπαϊκή Ένωση και Κίνα. Νομίζω ότι ένα νέο στοιχείο, τουλάχιστον στη δική μου είναι ότι η Κίνα είδε μια αλλαγή πολιτεύματος τα δύο τελευταία χρόνια. Ήταν μια κομμουνιστική αριστοκρατία Κίνα. Και τώρα έχουμε ένα σύστημα κομματικό αυτοκρατορικό το οποίο πλησιάζει τη δικτατορία όλο και περισσότερο καθημερινά. Αυτή είναι σημαντική αλλαγή. Νομίζω επίσης ότι η εξωτερική πολιτική της Κίνας ακολουθεί νέες οδούς. Να ρωτήσω λοιπόν ένα από τους εισηγητές που αναφέρθηκε στον Deng Xiaoping να μου πει κατά πόσο ακολουθεί την δική του εξωτερική πολιτική. όσον αφορά την επίδειξη δύναμη και το πότε γίνεται αυτό. Βλέπουμε ότι ο τωρινό ηγέτη δεν ξέρω κατά πόσο αυτό κάνει. Πρέπει να δούμε επίση το κατά πόσο αυτές οι διεθνείς αξίες, οι διεθνώς ισχύουσες αξίες που βρίσκονται και στις χάρτες του ΟΗΕ, κατά πόσο τις ασπάζεται και η Κίνα. Η Κίνα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους διασώτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο παρελθόν, τώρα έχει μια προσέγγιση διάρκεια βασίλευε για την Ευρώπη. Αυτό λοιπόν το ΣΥΝ 16 το σχέδιο είναι πραγματικά διχαστικό και συμφωνώ ότι η στάση κάποιων μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών νομίζω ακολουθούν μόνο τα δικά τους εθνικά συμφέροντα. Οπότε και αυτό είναι διχαστικό. Οπότε θα πρέπει να σταματήσουμε να άλλο κατηγορούμαστε και να καταλάβουμε επιτέλους ότι εδώ εκμεταλλεύονται αυτή την αναμία μας. Θα μπορούσαμε λοιπόν, θα έπρεπε μάλλον λοιπόν, να ακολουθήσουμε μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σόλτς, εξωματός της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω του εισηγητέ για τι παρουσιάσει του που βεβαίω μα έδωσαν μια ευκαιρία για άλλη μια φορά να ακούσουμε την ιστορική αναδρομή του σχέσεων μεταξύ ΕΕ και Κίνας. Αλλά ίσως θα πρέπει να εξετάσουμε ή να έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, μέχρι το 2030 και το θεματολόγιο του ΟΗΕ λείπουν 12 χρόνια. Οπότε θα πρέπει να έχουμε κάποιους κοινού στόχους και καθήκοντα για να δούμε ακριβώς τι κάνουμε για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους του 2030. Και αυτό βέβαια θα το κρίνει και θα το αποτιμήσει και ο τελευταίος πολίτης και στην Κίνα αλλά και στην Ένωση την Ευρωπαϊκή. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσο κατά πόσο θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα διεθνές, διεθνές σύστημα κανόνων και αξιών και κατά πόσο πρέπει να το εφαρμόσουμε. Το θέμα είναι λοιπόν το πώς εμείς θα ζούμε, θα παράγουμε και θα καταναλώνουμε ε, σε κάποια χρόνια. Και αυτά αφορά και την Ένωση, αλλά και την Κίνα, αλλά και τη ΣΥΠΑ και άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε μια νέα πραγματικότητα. Και νομίζω ότι η είσοδος της Κίνα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία την άλλαξε την ίδια την παγκοσμιοποιημένη οικονομία με νέες αντιφάσεις και προκλήσεις μπροστά μας που δεν είχαμε στο παρελθόν και που θα πρέπει με ενιαίο τρόπο στρατηγικά να αντιμετωπίσουμε. Θα έπρεπε λοιπόν να δούμε το θέμα του κατά πόσο αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες που υπάρχουν ώστε να συμβάλλουμε σε μια παραγωγική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ευχαριστώ. Και περνάμε στους τελευταίους δύο μιλητές από το ΕΛΚ και οι δύο Κούκαν. Ευχαριστώ. Οι εμπορικές σχέσεις ήταν τεταμένες. Ε, τελευταία ο επίσημος διαστρωμένος διάλογος ε, είναι περιορισμένος από την δική μας οπτική γωνία είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουμε ε, της, ε, την ανίσχυση του εμπορικού διαλόγου και είναι πολύ σημαντικό αν αυτός ενταχθεί αν αυτός ενταχθεί σε γενικότερα φόρουμ της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. Τι περιμένετε από τον, διάλογο, τον εμπορικό διάλογο στο μέλλον και τι στοιχεία θα πρέπει να εισάγουμε εμείς στην πολιτική μας ε, ε, την πολιτική των σχέσεων μας με την Κίνα έτσι ώστε να αποκλιμακωθούν. Ευχαριστώ κυρία Αντρικιέν. Έχω κλείσει τον κατάλογο των μιλητών, συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος ε, Λάινεν είπε ότι πρέπει να ξυπνήσουμε και νομίζω ότι ξυπνάμε ήδη. Ε, υπάρχει μια κινέζικη παροιμία που λέει ότι αν θέλει να γίνει πλούσιος χτίσει ένα δρόμο. Ε, μας ε, θυμίζει το ε, πρόγραμμα για την, τις ζώνες και του δρόμου της Κίνας. Ε, κάνει πολύ μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές αλλά και σε τεχνολογικές εταιρείες υψηλού επίπεδου. Αυτό έχει ανησυχήσει πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες. Χρειαζόμαστε μια κοινή εμπορική στατική για να αντιμετωπίσουμε την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται απαραίτητο ξένες ε, επενδύσεις, ξένες, άμεσες ξένες επενδύσεις. Αλλά χρειάζεται και ένας μηχανισμός επιλογής αυτών των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στρατηγικά σημαντικούς τομείς όπως η άμυνα, επικοινωνίες, ενέργεια, μεταφορές, τομείς από τους οποίους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ασφάλεια των πολιτών μας. Οι επενδύσεις και η άμεση, ο άμεσος ή έμεσος έλεγχος τους θα πρέπει να ε, βρεθεί στο μικροσκόπιο μας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη. Ο προστατευτισμός αυξάνεται και το εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες πλήττεται. Ε, σταθερές οικονομικές σχέσεις εξαρτώνται από αμοιβαιότητα οπωσδήποτε. Οπότε για να παίζουμε όλοι με τους ίδιους κανόνες η Κίνα θα πρέπει να ανοίξει την αγορά της στους ξένους επενδυτές με να βελτιώσει το ρυθμιστικό πλαίσιο, να προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα και λοιπά. Θα μπορούσαν οι ομιλητές να μου πούνε δύο λόγια για αυτό το θέμα. Um, Ευχαριστώ. Στόχος είναι να τελειώσουμε το αργότερο στις 4, οπότε έχουμε πέντε λεπτά μόνο. Στις 4 παρα 10, συγγνώμη, έχουμε πέντε λεπτά. Οπότε να ξεκινήσουμε ανάποδα.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 μειώσουμε τις διακρίσεις στην ε, εξωτερική εμπορική πολιτική της Κίνας. Το ερώτημα είναι χρειαζόμαστε μια βιομηχανική πολιτική αντίστοιχη της Κίνας. Δεν έχω απάντηση. Οι πολιτικοί μας ηγέτες πρέπει να το συζητήσουν. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Κίνα να γίνει σημαντικός παίκτη στους διεθνείς οργανισμούς μεταξύ αυτών και των ΠΟΕ. Θα πρέπει να καλέσουμε την Κίνα εκεί όπου διαμορφώνονται οι μελλοντικοί κανόνες τη παγκόσμιας διακυβέρνησης, για παράδειγμα τα διεθνή πρότυπα, και εκεί να έχει συμφέρον να εμπλακεί. Ε, αλλά θα πρέπει και η ίδια να μας το ζητήσει. Σε ό,τι αφορά την ομάδα 16 συν 1, ίσως είναι ένας τρόπος να διασκεδάσουμε τις υπόνοιες ότι πρόκειται για μια προσπάθεια διέρη και βασίλευε. Γι' αυτό το λόγο ίσως θα πρέπει να κάνουμε αυτές τις επενδύσεις στην, στην Νότια Ευρώπη. Υπάρχει ένα θέμα σύγκλησης μεταξύ της Κίνας και της Δύσης. Άλλοι Κάποιοι λένε ότι αυτή η σύγκληση δεν συμβαίνει. Ίσως είναι λίγο νωρίς να το πούμε. Αλλά η σύγκληση συνεχίζεται καθημερινά στον οικονομικό τομέα και θα συνεχιστεί. Αυτό είναι καλό και για την Κίνα και για μας. Η αντίφαση είναι ότι η Κίνα που αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πιστεύει πάρα πολύ στο μέλλον της. Ενώ η Ευρώπη που έχει όλες τις συνθήκες που χρειάζονται για ένα λαμπρό μέλλον δεν είναι τόσο αισιόδοξη πάντοτε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αισιόδοξοι για το μέλλον μας. Γιατί αυτό θα μας έδινε και μοχλοπίεση στη σχέση μας με την Κίνα. Τώρα, η Κίνα θα προχωρήσει με τα ρυθμίσεις της. Ο πρόεδρος θα καταφέρει. Θα πρέπει να πούμε στην Κίνα ότι είναι πολύ σημαντικό να ελοπίσει τη δεσμεύση της. Αυτό πρέπει να της το καταστήσουμε σαφές. Η έλλειψη αμοιβαιότητας ε, δημιουργεί προβλήματα. Και σε αυτό το στάδιο υπάρχει έλλειψη αμοιβαιότητα. Η Κίνα θα πρέπει να προχωρήσει σε πιο βαθίε μεταρρυθμίσει και να ανοίξει την οικονομία τη περισσότερο. Η... η άνοδος της Κίνας ε, είναι αναπόφευκτη. Δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι κοινοτοπία αλλά είναι πραγματικότητα. Μια δύναμη Κίνα όμως θα ήταν κάτι πολύ κακό για όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να εμπλέξουμε την Κίνα στον δρόμο της ανάπτυξης μαζί μας. Και δεν θα πρέπει να έχουμε... Ε, να τρομοκρατούμαστε. Ας προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία αυτό το περίπλοκο πρόβλημα της Κίνας. Όταν οι δικές μας απόψεις για την Κίνα είναι πολύ ακραίες, οι Κινέζοι, αυτό ξυπνάει το φόβο των Κινέζων ότι υπάρχει μια διεθνή συνωμοσία εναντίον τους και αυτό επηρεάζει τις επιχειρήσεις και το διάλογο. Θα πρέπει οπωσδήποτε ο διάλογος να συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε θέματα αριθμιστικού πλαισίου. Ο προτελευταίος ομιλητής μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις. Η Κίνα έχει ευθύνη να ενημερώνει πολύ περισσότερο τη Δύση για το πολιτικό τη σύστημα ε, και τις αλλαγές τις οποίες επιφέρει, γιατί αυτά φοβίζουν τη Δύση. Και όπως είπε ο τελευταίος ομιλητής, ε, αν εστιάσουμε στο θέμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τότε βέβαια η δράξει της ε, Κίνας είναι απολύτως απαραίτητε, Είναι πολύ σημαντικές για, για την επιτυχία των στόχων αυτών. Πέρσι είδαμε πολύ πιο αυστηρή εφαρμογή των περιβαλλοντικών καμονών, οριζόντια, ε, και τα τελευταία χρόνια η Κίνα επενδύει όσο περισσότερο οποιαδήποτε άλλη χώρα σε ε, ανανόσιμες πηγές ενέργειας και αυτό βοηθάει και τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Αυτές είναι οι εξέλιξες ό,τι αφορά το περιβάλλον στην Κίνα. Η, ε, συμπέρασμα η Ευρώπη θα πρέπει να εμπιστευτεί την οικονομία της, να δει το μέλλον της με αισιοδοξία, γιατί αυτό της δίνει μοχλοπίεσης. Η Κίνα είναι σημαντική και για τις ευρωπαϊκές εταιρείε θα γίνει ακόμα πιο σημαντική στο μέλλον. Οπότε ας συνεχίσουμε τον βαθύ διάλογο με την Κίνα ε, και ιδιαίτερα για θέματα ρυθμιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. now, Mr. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάντερ Πούτεν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βάντερ αλλά και άλλοι ομιλητές μίλησαν για νέες συζητήσεις για τη στρατηγική μας για την Κίνα. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μου σε δηλαδή τις εξελίξεις στη χάραξη τη νέα πολιτική. Το πρώτο συστατικό αυτή της νέα στρατηγική. Καταρχά θα πρέπει να παρουσιάσει μια σαφή εικόνα του πώ θα δείχνει το νέο παγκόσμιο σύστημα. Δηλαδή θα αλλάξει το status quo και το νέο σύστημα θα εξελιχθεί, θα διδραματίζει και σημαντικό ρόλο η Κίνα. Mm. Αλλά βέβαια αυτό θέτει το ζήτημα το ποιο θα είναι, ποιος θα είναι και ο ρόλος της Ένωσης μαζί με τον ρόλο της Κίνας βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τη μέγιστη δυνατή ευρωπαϊκή επιρροή διατηρώντας ταυτόχρονα τις ευρωπαϊκές αξίες παγκοσμίω. Βέβαια θα είναι πιο λεπτομερής αυτή η νέα στρατηγική από αυτό που λέω τώρα. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορά διλήμματα γιατί έδειξε εδώ η συζήτηση ότι αν επικεντρωθούμε μόνο σε διάφορα υποθέματα, δεν θα είναι σαφές το ποια είναι η συνολική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγάλα διλήμματα πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η επιλογή μεταξύ των ανθρωπίνων πούμε, δικαιωμάτων και συναφών αξιών και τα οικονομικά και πολιτικά ενδιαφέροντα και συμφέροντα της Ένωσης από την άλλη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία θα εφαρμόζονται και τα οποία θα μας καθοδηγούν για το πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτά τα διλήμματα. Οι επενδύσεις και η αξιολόγησή τους. Τι γίνεται επίσης με την Ταϊβάν. και η φύση της σχέσης μας. Γιατί έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις για την Κίνα. Αν θέλουμε όμως να μετατραπούν σε μια ενιαία ιδέα και αντίληψη για την Κίνα, τότε και αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Επίσης θα πρέπει να βρούμε ένα νέο αφήγημα για το πώς αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις επενδύσεις παγκοσμίω. Είδαμε ότι και να έχει το δικό της αφήγημα για τις επενδύσεις, το οποίο σχετίζεται άμεσα με τον δρόμο του μεταξιού και την πρωτοβουλία αυτή και φαίνεται να ελκύει πολλούς παγκοσμίω. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο το αφήγημά μας δεν ήταν μέχρι τώρα επαρκώς επιτυχές και κατά συνέπεια θα πρέπει να βρούμε άλλο αφήγημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια σαφέστερη προσέγγιση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς εμείς προσεγγίζουμε το θέμα της ανάπτυξης γενικότερα στο 21ο αιώνα. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι σε πολλές χώρες του κόσμου εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ενδεχομένω και εντός Ένωσης για περισσότερη οικονομική ανάπτυξη και εκεί θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι έχει να προσφέρει η Κίνα και ο δρόμος του μεταξύ εδώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα ήταν λοιπόν καλό από στρατηγική σκοπιά για την Ευρώπη να προβληθεί η ιδέα για μια πρώτα σε σχέση με τη μορφή που θα έχει αυτός ο δρόμος του μεταξιού, μιας και αφορά αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι το ίδιο με το BRI που είναι καθαρά κινέζικη πρωτοβουλία και που συμβαδίζει με την πρωτοβουλία για το δρόμο του μεταξύ. Αυτά από μένα πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και πρόεδρος. Ο κύριος Βάντεφελ πέντε λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δύο σύντομα σχόλια για τις επενδύσεις. Ναι, μας λείπουν ακόμα στοιχεία σε σχέση με τις επενδύσεις. Για τις διμερείς σχέσεις, επίσης, να κάνω δύο σύντομα σχόλια. Δεν έχουμε μόνο τις επενδυτικές συμφωνίες, αλλά και το θέμα των φραγμών, των εμπορικών που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Επίσης, ενδεχομένως να μην συναφθεί καθόλου ή να μην ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία επενδυτική. Για τον ανταγωνισμό τώρα. Είχαμε πολλές παρατηρήσεις. Καταρχά το ζήτημα του κατά πόσο η δύναμη της Κίνας οφείλεται σε ευρωπαϊκές πολιτικές. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Αναφερθήκαμε στο 16 1. Το 16 1 είναι ένα αποτέλεσμα κάποιων μη αποτελεσματικών ευρωπαϊκών πολιτικών που το εκμεταλλεύεται η Κίνα αυτό και προκλεί κάποιους πολιτικούς διχασμούς τους οποίους εκμεταλλεύεται πολιτικά και οικονομικά η Κίνα. Βεβαίως και οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν και στους ιδιαίτερες σχέσεις με την Κίνα και παραβλέπουμε καμιά φορά το γενικότερο ευρωπαϊκό συμφέρον. Και στις πρωτεύουσες θα πρέπει να το σκεφτούν σοβαρά αυτό. Επίσης, να μην είμαστε αφελείς σε σχέση με την πολιτική ταύτιση Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αν δούμε τι γίνεται, ας πούμε, στις ε, διατυπώσεις ή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται, ε, σε κάποια θέματα υπάρχουν κάποιες ε, συγκλήσεις, αλλά όχι. Και να μην ξεχνάμε επίσης ότι αυτό το κοινωνικό πρότυπο είναι αρκετά ελκυστικό για πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό να το θυμόμαστε. Και υπάρχει και συγκεκριμένο λόγος γι' αυτό. Επειδή η οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια της Κίνας είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οπότε, αν το δει κανείς απ' έξω, είναι αποτελεσματικό το μοντέλο τους. Βέβαια, αφού και ο κ. σε κάποιες αλλαγές που έγιναν. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι λιγότεροι φοιτητέ πηγαίνουν στην Κίνα επειδή δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ, facebook, twitter κλπ. Θα πρέπει λοιπόν να το κοιτάξουμε αυτό, να δούμε κατά πόσο υπάρχουν περιορισμοί σε αυτά τα θέματα, τουλάχιστον σε σχέση με τους πολίτες της Δύσης. Και το λέω αυτό απλά και μόνο παράδειγμα. Επίσης, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός μας ή μάλλον σχεδιασμός της Κίνας είναι αναπόσπαστο τμήμα της επιτυχίας τους. Τώρα όμως θα πρέπει να δούμε α, τι θα γίνει ας πούμε ο ηγέτης τους, ο Σιζι ε, πάθει ανακοπή καρδιάς, πάθει καρδιακό. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ε, οπότε θα πρέπει να έχουμε και εναλλακτικέ. Επίσης μιλάμε για κινέζικα χρήματα που είναι πακτολός. Αυτό δεν είναι το μοναδικό στοιχείο επιτυχίας στην Ινδονησία είπαν ότι δεν είναι και τόσο επιθυμητά, δεν είναι και τόσο λογιστικά, είπαν στην Ινδονησία, επειδή σημαίνει και επιρροή, οπότε δεν το θέλουμε αυτό. Οπότε το χρήμα από μόνο του δεν κυριαρχεί. Οπότε εμεί ω Ένωση δεν πρέπει να ανταγωνιζόμαστε του κοινού σε αυτό το επίπεδο, το οικονομικό δηλαδή. Θα πρέπει να δούμε πώ πραγματικά θα μπορούσαμε να το συμπληρώσουμε, αλλά να χρησιμοποιήσουμε και άλλες ε, μεθόδους, άλλες πηγέ, α πούμε εκπαίδευση κτλ, ώστε να έχουμε ένα αποτέλεσμα. Οι κινέζικε πολιτικές και επιρροή του το lobbying στην Ευρώπη. Είναι δημόσιες σχέσεις και έξυπνη διπλωματία. Δεν θέλω όμως να επιστρέφω σε αυτό σε βάθος, γιατί αρκεί να σας πω το εξής. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε αντίστοιχα αυτό που κάνουν οι Κινέζοι στην Κίνα. Οπότε θα πρέπει γενικότερα να δούμε το ευρωπαϊκό συμφέρον. Δεν θα πρέπει να ασχολούμαστε συνέχεια με τις είπα και το τι κάνουν. Εντάξει, σημαντικό είναι. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τα χαμηλά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως Ευρωπαίοι Υπάρχουν βέβαια κάποια κοινά συμφέροντα με τις ΙΠΑ σε θέματα εμπορίου, επενδύσεων κτλ. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στη σχέση μας με την Κίνα δεν έχει αλλάξει τίποτα λόγω Τραμπ. Υπάρχει έλλειψη αμοιβαιότητας όσον αφορά τις σχέσεις τις επενδυτικές, έχουμε πρακτικές αθέμητες ακόμα, έχουμε αποκλίνουσες επίσης απόψεις, ε, συγγνώμη αξίες Αποκαλύπτουν όλο το φάσμα σχέσεων και αν μπορούμε να πετύχουμε κάποια σύγκληση στο επιχειρηματικό κομμάτι θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του η, η οποιαδήποτε επιτυχία σε αυτό το κομμάτι την στάση των Κινέζων και τη δικιά τους πολιτική. ΠΟΕ τώρα. Δεν υπάρχει απόλυτη ταύτιση και λόγω Τραμπ δεν θα πρέπει εμεί να δώσουμε υπερβολικό βάρο στην ε, Κίνα σε αυτή την περίπτωση. Στα πλαίσια του ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, του ε, τρει εισηγητέ μα. Σα ευχαριστώ που ήρθατε. Έχει αποσυνδεθεί και ο εισηγητής μα από το Πεκίνο. Ευχαριστώ λοιπόν για τις εισηγήσεις σα. Μας μπέλετε μήπως θέλει να μα πει κάποια σχόλια τελικά. Έχει τον τελευταίο λόγο. Παρακαλώ. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η ακρόαση καταδεικνύει ότι θα πρέπει να έχουμε περισσότερη συνεργασία, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα από κοινού, κοινοβούλιο, συμβούλιο, κομισιόν και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει γιατί πρέπει να κάνουμε πιο πολλά και περισσότερο σε βάθος ώστε πραγματικά να μειώσουμε ή να εξαλείψουμε οποιαδήποτε ένταση ή αδυναμία που υπάρχει μεταξύ των δύο μερών αυτή τη στιγμή. Πρέπει επίση να διατηρήσουμε την ενότητά μας. Το Ινστιτούτο Μακάρθη έκανε κάποιες μελέτες από αυτού και ο κ. Βάντεφελ νομίζω το ανέφερε προηγουμένως και χαίρομαι για αυτές τις μελέτες που αναφέρθηκε ο κ. Βαντεπούτεν από την Χάγη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για αυτή την επιστημονική συμβολή στην ε, δουλειά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Είστε επανειδήν. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Uh, Ωραία, συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει. Γι' αυτό και θα πρότεινα να περάσουμε αμέσω στο σημείο 18, σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση Κίνα, έπειτα από την ακρόαση που μόλι διοργανώσαμε